Good afternoon. Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μου. Καταρχήν να σας καλωσορίσω όλους θερμότατα σε αυτή τη συνεδρία σε συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην νέα κοινοβουλευτική θητεία. Θα προεδρεύσω στα πορτογαλικά, γι' αυτό ετοιμαστείτε. Για αλλαγή. Και είναι και ωραία γλώσσα στο κάτω-κάτω για τα πορτογαλικά. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι η Προεδρία στη συνεδρίαση την ασκεί προσωρινά ένας από τους ε, απερχόμενους αντιπροέδρους ε, με βάση την τάξη. Καταρχήν, ε, ο ένας απερχόμενος πρόεδρος δεν είναι τακτικό μέλος, η Τανίδα Χούμπνερ, την καλωσορίζω παρόλα αυτά στην Επιτροπή, οπότε να πω και σε μένα Ω αντιπρόεδρο απερχόμενο της Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων να ασκήσω την Προεδρία προσωρινά μέχρι την εκλογή του Προέδρου και να κηρύξω την έναρξη της συνεδρίασής μας. Είναι γνωστός ο σκοπός αυτής της συνεδρίασης. Είναι η σύσταση του Προεδρίου της Επιτροπής ΑΦΚΟ με τις αρχαιρεσίες του Προέδρου και των Αντιπροέδρων. Και θα εκλέξουμε όπως είναι φυσικό πρώτα τον πρόεδρο και κατόπιν το κάθε αντιπρόεδρο ξεχωριστά. Δικαιούνται να ψηφίσουν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής και κάποια αναπληρωματικά μέλη που αντικαθιστούν τακτικά μέλη εφόσον ε, οι πολιτικές ομάδες έχουν ανακοινώσει τις αντικαταστάσεις. Ε, έχω τον εξής κατάλογο για ανα, αντικαταστάσεις. Ο κύριο Βίλαντ αντικαθιστά την κυρία... ή μάλλον η κυρία Χίμπρερ μάλλον αντικαθιστά τον κύριο Βίλαντ. Μπενιφέ Ρίτσαρ Κόρμπετ. τζειμ Wells αντικαθιστά τον Ρόμπερτ Λόφ. Η Κίνκα Γκόλ αντικαθιστά τον Λοράν Ζορτζι Βίντς και ο Γκέρτ Μπουρζουά αντικαθιστά τον Ντάνιελ Χάνον. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλες αντικαταστάσεις. Πρέπει να δηλωθούν τώρα. να ενημερωθεί το Προεδρείο πριν τις εκλογές. Η Ντανούτα Χίμπνερ, εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Σαν Σάιμον, ποιον αντικαθιστώ. Καλά στο σημειώνουμε. Τον Παύλο Ραζέλ αντικαθιστάτε, μάλιστα. Έχουμε εξακριβώσει την απαρτία για να είναι έγκυρη η ψηφοφορία και οι εκλογές. Ο Ασκόν την Προεδρία ερωτά την Ομίγυρη. Υπάρχουν προτάσεις για υποψηφιότητες για την Προεδρία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Ποιος ήθελε το λόγο. Φαντάζομαι η Ντανούτα Χούμπνερ έχει να κάνει μια πρόταση. Θα ήθελα εκ μέρους του ΕΛΚ να προτείνω τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Αντώνιο Ταγιάννη, για την προεδρία της Επιτροπής ΑΦΚΟ, της Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων. Μάλιστα. Ευχαριστώ για την πρόταση. Μας ε, εξέπληξε όλους αυτή η πρόταση. Ερωτώ λοιπόν τον υποψήφιο αν δέχεται την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ και το αποδέχομαι κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα, ευχαριστούμε και εμείς. Φαντάζομαι ότι έχει κάνει τη δήλωση του Ποθενέσχες τη δήλωση με βάση τον δεντολογικό κώδικα, οπότε μπορούμε να περάσουμε στην εκλογή. Υπάρχει άλλος υποψήφιος καταρχήν για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Όχι, οπότε προτείνω να ψηφίσουμε δι και να επικυρώσουμε την εκλογή του το στην Προεδρία. Μάλιστα. Εκλέγεται ο κύριος Σταγιάννη και τον παρακαλώ να έρθει στο Προεδρείο και να λάβει τη θέση του Προέδρου. is not perfect. Είναι και άπτυστα τα πορτογαλικά μου. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την εκλογή των αντιπροέδρων. Υπενθυμίζω στα μέλη της Επιτροπής μας πως δυνάμει το άρθρο 213 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο Προεδρείο κάθε Επιτροπής η σύνθεση του Κοινοβουλίου με την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. Ε, άρα λοιπόν δεν μπορεί ούτε να είναι του αυτού φίλου ούτε προερχόμενοι από το ίδιο κράτος μέλος ή αντιπρόεδροι. Και παρακαλώ να γίνει σεβαστό αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε κάποια παρατήρηση εν προκειμένου. Κυρία Φίμπνες. Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω να κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα για τους συντονιστές, ώστε να συζητήσουμε τα θέματα επιλογής υποψηφίων αντιπροέδρων, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε με επιτυχία τις εκλογές αντιπροέδρων. Καλώς, λοιπόν, παραχωρώ πέντε λεπτά διακοπή για τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. δεν έχουμε λόγο να κρύψουμε. Έχει πια προχωρήσει τόσο πολύ η κατάσταση στο κοινοβούλιο που δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Πέντε λεπτά διάλειμμα ή όποτε μπορέσετε να τελειώσετε τη δουλειά σας. Are you ready? Yes, uh, Mrs. Yes, Chair, I would like to announce on behalf of all my colleagues that... Εκ μέρους των συναδέλφων θα ήθελα να ανακοινώσω, κύριε Πρόεδρε, πως εξευρέθη, πως δεν εξευρέθη συμφωνία και άρα θα πρέπει να αναβληθεί μέχρι Δευτέρας η ψηφοφορία για τον πρώτο πρόεδρο, αλλά για να ολοκληρωθεί η συγκρότηση πρέπει να ψηφιστεί πρώτος αντιπρόεδρος ακόμη της Επιτροπής μας. Επομένως, είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε με την ψηφοφορία για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Μάλιστα. Δηλαδή, οι συντονιστέ προτείνουν να ψηφιστεί ο πρώτο αντιπρόεδρο και μέχρι Δευτέρα στο Στρασβούργο να αναβληθεί η ψηφοφορία για τον τρίτο τέταρτο αντιπρόεδρο. Yeah. Yes, yes, Vi informato che è necessario. Ενημέρωσα ότι απαιτείται να έχουμε τουλάχιστον μία γυναίκα μεταξύ των τεσσάρων αντιπροέδρων. Αν εκλεγεί σήμερα λοιπόν ως πρώτος αντιπρόεδρος άντρα συνάδελφος, για να εξαρτήτως των πολιτικών προβλημάτων και δυσκολιών, υπάρχει ζήτημα και ισορροπίας φύλων Να το ξέρετε. Οι σοσιαλιστές δημοκράτες μου λέγεται πως θα ήθελα να καταθέσουν υποψηφιότητα γυναίκας για αντιπρόεδρο. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ. Όντως οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες με χαρά υποβάλλει την υποψηφιότητα της κυρίας Γκαμπριέλ Μπίσοφ για τη θέση της πρώτης αντιπρόεδρου. Και αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό ακόμα, να σας ε, συγχαρώ επ' ευκαιρία για την εκλογή σας, Πρόεδρε. Και η ομάδα μας είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει ως πρόεδρο της Επιτροπής ΑΦΚΟ ένα πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά για μια ισχυρότερη και πιο ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Please. Haluaisin ehdottaa ID-ryhmän puolesta ensimmäiseksi varapuheenjohtaja. ευχαριστώ. Θα ήθελα να προτείνω τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου, της πρώτης αντιπροέδρου, την κυρία Άνεμαν, η οποία έχει χρόνια υπηρετεί στην Επιτροπή αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να είναι δυνατόν να ακουστούν όλες οι φωνές, γιατί έχουν καταψηφιστεί πολλές φορές γυναίκες εδώ. Ναι, βεβαίως. Θα ήταν καλό να γίνεται και γραπτός και μυστική η ψηφοφορία. Ωραία, λοιπόν, έχουμε την υποψήφια. Δέχεστε την υποψηφιότητα αυτή. Ευχαριστώ πολύ και επιτρέψτε μου να συστηθώ. Δέχομαι βέβαια την ε, υποψηφιότητα. Είμαι νέα βουλευτής, αλλά ασχολούμαι χρόνια με την ευρωπαϊκή πολιτική. Χρόνια πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αντιπρόεδρος του Φεντεραλιστικού Κινήματος της Γερμανίας, ε, αγώνιζομαι χρόνια για το φεντεραλισμό στην Ευρώπη και είχα και τη θέση του μόνιμου παρατηρητή στην ε, Στακτική Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης. Ελπίζω λοιπόν ότι θα με υποστηρίξετε. Εσείς παρακαλώ δέξτε την υποψηφιότητά σας. Πρόεδρε, ναι, σας πω γιατί. Οι διαπραγματεύσει μεταξύ διαφόρων ε, ομάδων γενικών γραμματέων, δηλαδή πριν από την ε, ανάθεση καθηκόντων σε πρόεδρο και την πρόεδρου της Επιτροπής, έδειχναν ότι ίσως να προκύψει πρώτος αντιπρόεδρος της ΙΝΤΕ στην ΑΦΚΟ και είπα σε αυτήν την περίπτωση μπορώ να δεχθώ εάν η ομάδα μου με υποστηρίζει. Ακούω όμως σφήμες πως το σύστημα DONT που είναι και ο λόγος υπέρ της αυτού του εγγράφου δεν εφαρμόζεται πλέον. Προέρχομαι από το Βέλγιο, τη χώρα που εφήβρε το κορδόν σανιτέρ. 35 χρόνια στο Βέλγιο, στην πολιτική ζωή, είδα κορδόν σανιτέρ. Αλλά δεν είδα αυτό να εφαρμόζεται ποτέ στην διοίκηση του Κοινοβουλίου. Μάλλον πρώτη φορά στην ιστορία, στη δημοκρατία των ανθρώπων και την ιστορία της δημοκρατίας των ανθρώπων. Βλέπουμε αυτό να συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λυπούμε βαθύτατα. Αλλά συνεχίζει να υπάρχει αυτό το έγγραφο και ίσως να υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία που είστε, που φαίνεται αποφασισμένη να ρίξετε πάνω στο κοινοβούλιο, να δει και μια εξαίρεση την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Είμαι χρόνια μέλος της Επιτροπής δεν είχα ποτέ προκλητικές ε, τοποθετήσεις ή στάση, πάντα ε, επιφυλακτικός, συνετός, μετριοπαθής, ακόμα και όταν επέκνα πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα κάνετε το ίδιο πράγμα στην ε, ΑΦΚΟ, όπως συνέβη με τις άλλες επιτροπές ή την Ολομέλεια. Υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες που έχουν ψηφίσει για την ομάδα μου και άρα ή θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαχείριση του Κοινοβουλίου ή θα αποκλειστούν όπως συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια ή όπως γίνεται αυτή τη στιγμή και σε άλλες επιτροπές. Παρακαλώ μην το πράξετε και στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ιδέαλος για πέντε χρόνια. 21 εκατομμύρια πολίτες και πολλοί ήταν Ιταλοί μεταξύ αυτών κύριε Πρόεδρε θα δουν ένα κοινοβούλιο με παραμορφωμένη εικόνα Ίσως η Επιτροπή Σταματικών Υποθέσεων είναι και συμβολικά μια πολύ καλή ευκαιρία να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, αξιοποιήστε αυτή την ευκαιρία ώστε τα 21 εκατομμύρια των μελών της ΕΔ να μην αποκλειστούν. Δεν αποκλείεται εμένα, δεν αποκλείεται την ομάδα ΕΔ, αλλά τους πολίτες τα 21 εκατομμύρια. Μην το κάνετε λοιπόν. Καλά. Και ενώ ετοιμάζονται τα ψηφοδέλτια για την ψηφοφορία. No, βοηθάμε με con la scheda. καρτάσιο, cartaceo. Ho chiesto voto cartaceo. καρτάσιο. Βαλκούνος... Έχει κανείς αντίρρηση στο να γίνει ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Σε, me si può fare... Πρόεδρε, μπορεί να γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία μυστική, όπως πράξαμε και στο Στρασβούργο. Eh? Ε, μα είναι αποφάση του Πρόεδρου, να ξέρετε. Αν δεν ζητεί κανεί ψηφοφορία επί χάρτου, με ψηφοδέλτιο, τότε μπορούμε να κάνουμε ψηφοφορία ηλεκτρονική. Εάν ζητάτε όμως επί χάρτου, με ψηφοδέλτιο, παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ψηφίσουμε με ψηφοδέλτια σε χαρτί. Secret secret is on the secret, Paper yes, is on the... I think paper is secret. Yes, but electronic too. Pas, pas l'obligé, parce que

Ε, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μυστικότητα, η ηλεκτρονική ψηφοφορία την ε, εξασφαλίζει. Το κάναμε και σε άλλες επιτροπές. Για τη μυστικότητα μας καλύπτει και η ηλεκτρονική ψηφοφορία, εκτός αν για άλλους λόγους θέλει κανείς ψηφοδέλτια. Αν συμφωνούν όλοι, δεν έχω αντίρρηση, κανένα πρόβλημα. Εάν συμφωνείτε όλοι. Αν όμως μας ζητούν αυτοί ψηφοφορία επί χάρτου δεν μπορώ να το αρνηθώ. Όχι, η απόφαση είναι του Πρόεδρου. Ε, ένα σχόλιο μόνο. Δεν νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε με ψηφοδέλτια. Αυτό που ε, απαιτείται είναι η μυστική ψηφοφορία, αλλά και η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι μυστική. Δεν υπάρχει λοιπόν ε, λόγος να ψηφίσουμε με ψηφοδέλτια. Η μόνη υποχρέωση που προβλέπει ο κανονισμό είναι να είναι μυστική ψηφοφορία. Αλλά ο πρόεδρο θα το αποφασίσει αν η μυστική ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά ή με ψηφοδέλτια. Ναι, ναι, όλα αυτά ο πρόεδρο θα το αποφασίσει. Απλώ λέω ότι η νομική υποχρέωση αφορά τη μυστικότητα, όχι το υπόθεμα. Ναι, ναι, είναι καθήκον του Προέδρου να δεχθεί την απόφαση της πλειοψηφίας και να προστατεύσει τη μειοψηφία για να μην μου πει κανείς ότι έχω κάνει κάτι που βλάπτει την ψηφία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι καλύτερο να ψηφίσουμε με ψηφοδελτία σε χαρτί. Α Ας ορίσουμε ψηφολέκτης λοιπόν. estraggono i nomi degli scrutatori. Βάζω με λαχνό τα ονόματα των ψηφολεκτών. Γκονσάλες Πόνς. Μποζελάγκερ. Εσείς οι δύο ψηφολέκτες.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 Sulla scheda ci sono i nomi dei due candidati, bisogna metterla. Στο ψηφοδέλτιο λοιπόν έχετε τα ονόματα των δύο υποψηφίων, θα βάλετε το στα, σήμα του Σταυρού δίπλα στο όνομα του ενός από τους δύο και μετά καταθέτετε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, υπογράφοντας βεβαίως. Um, if... Μπορείτε να μας διευκρινίσετε εάν εκλέγουμε σήμερα Προεδρείο και άρα θεωρείται ότι πλέον θα έχει συγκροτηθεί η ΑΦΚΟ και άρα θα έχουμε δύο άντρες μέλη, δεν παραβιάζονται εκεί οι σχετικές διατάξει του κανονισμού, εάν εκλεγεί άντρας. Ο Πρόεδρος. Εκλέγουμε πρώτο αντιπρόεδρο. οι συντονιστές ε, κατέληξαν στη συμφωνία να ψηφιστούν στις 3 ε, ε, ο τρίτος και ο τέταρτος αντιπρόεδρος την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ο πρώτος αντιπρόεδρος, εφόσον εκλεγεί άντρα, ο τρίτος και ο τέταρτος θα πρέπει να είναι γυναίκες. Εάν όχι, τότε Εάν δηλαδή εκλεγεί γυναίκα στη θέση του πρώτου του Προέδρου, τότε δεν πειράζει τι θα γίνει στη συνέχεια. Ένας από τους τέσσερις δηλαδή τουλάχιστον πρέπει να είναι γυναίκα και εφόσον είναι άντρα ο πρόεδρος. Εάν εκλεγεί γυναίκα δεν θα χρειαστεί θέση άλλης γυναίκας στο Προεδρείο. Βεβαίω και μπορεί να εκλεγεί άλλη γυναίκα, αλλά όχι υποχρεωτικά. Εάν όμως εκλεγεί άντρα σήμερα, τότε οπωσδήποτε μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι γυναίκα από τους ε, τρίτο και τέταρτο αντιπρόεδρο που θα εκλεγούν στο Στρασβούργο. Please. I can add to what you have said. Θα ήθελα να προσθέσω αυτά που είπατε κύριε Πρόεδρε, ότι η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία ID, επαναλαμβάνω, η ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία είναι ανοιχτή. Εγώ, συντονιστή τη ομάδα ID, είμαι πρόθυμο να συζητήσουμε οτιδήποτε και ενδεχομένω να αντικατασταθώ από τη συνάδελφο για το Αυτό σε απάντηση της δικής σας ερώτησης προηγουμένως. Εμείς δεν επιβάλλουμε κανέναν άνδρα, δεν προτιμούμε άνδρα. Είμαστε ανοιχτοί στις συζητήσεις που πρότεινε για τη Δευτέρα κυρία Χιούμπνερ. δεν είπε κανεί ότι προσπαθείτε να επιβάλλετε παρουσία άντρα στο Προεδρείο. Απλώ ο συνάδελφο ρώτησε αν αυτό, σύμφωνα με του κανόνε, σημαίνει πω εκλέγονται και οι λοιποί αντιπρόεδροι. Όχι. Για τη συγκρότηση αρκεί να εκλεγεί ένα αντιπρόεδρο. Αν εκλεγείτε εσεί, για τους, για τους άλλους τρεις αντιπροέδρους, αυτούς που ακολουθούν δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα. Εάν εκλεγεί η κυρία Μπίσοπ, οι τρεις λοιποί μπορούν να είναι άντρες ή γυναίκες. Αφού ο πρόεδρος είναι άντρας λοιπόν, το επαναλαμβάνω, από τους τρεις αντιπροέδρους, μία τουλάχιστον πρέπει να είναι γυναίκα. team against Proclamo i risultati per l'elezione del primo Ανακοινώνω τα αποτελέσματα για την εκλογή πρώτου αντιπροέδρου. Εψήφισαν 26. Η κυρία Μπίσοπ έλαβε 17 ψήφους, ο κύριος Άνεμανς 8, ένα λευκό. Εγκλέγεται πρώτη αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΑΦΚΟ η κυρία Μπίσοπ και την καλώ στο Προεδρείο. Συγχαρητήρια. La riunione, la prossima riunione... Η προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής μας κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα το βράδυ στο Στρασβούργο με ημερήσια διάταξη την εκλογή των τριών αντιπροέδρων. αφού εξελέγει πρώτη πρόεδρος γυναίκα, δεν απαιτείται πλέον να υπάρχουν άλλες γυναίκες ως υποψήφοι. Δυνατό βέβαια πάντα, αλλά όχι απαραίτητο. Δυνάμει του κανονισμού. Έχει καλυφθεί ο όρος της εκπροσώπησης των φίλων. Έχετε λάβει και το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων μέχρι το πέρας του έτους. Εάν δεν έχετε αντίρρηση το εγκρίνουμε. Και μπορούμε να πάμε με την Αντιπρόεδρο Μπίσοπ για τη φωτογράφηση. Και τα ξαναλέμε στο Στρασβούργο τη Δευτέρα. Κυρία Μπίσοπ. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε επικοδομητικά και να βάλουμε καλές προδιαγραφές και στην Επιτροπή για ένα καλό κοινοβούλιο και καλή διοργανική ισορροπία. Ναι, και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Μπίσοπ, αλλά και τον έτερο υποψήφιο. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Θα ακολουθήσω τη στάση που είχα και ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Κάθε βουλευτής εκπροσωπεί ψηφοφόρους, κάθε βουλευτής θα τύχει του σεβασμού μου, κάθε βουλευτής θα έχει την ίδια αξία με τον έτερο βουλευτή. Η πόρτα του γραφείου μου είναι πάντα ανοιχτή, για κάθε αίτημα, για κάθε πρόταση, θα είμαι στη θέση σας πάντα. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το ειδικό βάρος του Κοινοβουλίου. Πολλές φορές και ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχα πει πως είναι καλό να αγωνιζόμαστε για να εξασφαλιστεί και το δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. είμαστε το μόνο Κοινοβούλιο που δεν έχει στον κόσμο ε, δικαίωμα πρωτοβουλίας. Πολλά πρέπει να κάνουμε λοιπόν και εμείς και ως Επιτροπή ΑΦΚΟ βεβαίως. Από αυτήν την έποψη λοιπόν ελπίζω να συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες. Αν θέλουμε ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχυρό πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα για το Κοινοβούλιο και εξονόματος των Ευρωπαίων πολιτών να καταθέτουμε νομοθετικές προτάσεις ε, και να μην εξαρτώμαστε μόνο από τις προτάσεις της Επιτροπής, βεβαίως και έρευνες και τα αλλά και άλλα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν, που είναι το ε, Brexit οπωσδήποτε, αλλά πολύ πιο λεπτό θέμα. Πάντως θέλω το, η Επιτροπή μας να καταστεί ε, πρωταγωνίστρια της επιδίωξης για μια εκπροσώπηση πολύ πιο ουσιαστική του εισψήφου των πολιτών που ξέρουμε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την εξέλιξη των πραγμάτων. Πρέπει να τους δώσουμε πιο πολλές απαντήσεις και η εξουσία αυτή για το Κοινοβούλιο είναι η καλύτερη απάντηση που μπορούμε να προσφέρουμε στον πολίτη. Είμαι διτεθειμένο να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Είμαι στη διάθεση όλων των συναδέλφων που μπορεί να έχουν την ίδια ιδέα με μένα, την ίδια έποψη και διαφορετική τελείω. Πάντως θα κάνω ό,τι πρέπει από το χέρι μου, θα αγωνιστώ όσο μπορώ, ώστε η απόσταση μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων να μειώνεται. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ε, διαβεβαιώ για την απόλυτη διάθεση για συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.